και τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα. Ε, θα ενημερώνουμε συνεχώς το Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, κύριε Τεχόχτ. Έχω λάβει δύο ψηφίσματα. Ε, το ένα είναι από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και το άλλο από την ομάδα των Πρασίνων και της Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.30. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη σας λέγω ότι δεν έχει ζητηθεί να ε, ψηφιστούν εκθέσεις που πρόκειται να διαδοθούν μέχρι τις 5.30 και θεωρούνται εγκεκριμένες. Το επόμενο θέμα ερώτηση με έτοιμα προφορικής απάντησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εμπορικέ Σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Ταϊβάν. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στο συνάδελφο κύριο Κασπάρη για πέντε λεπτά, συντάκτη της ερώτηση. Παρακαλώ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Το συνολικό ύψο διμερίσεω εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ταϊβάν ξεπέρασε τα 40 δισεκατομμύρια το 2011 και πέρυσι ε, εντάθηκαν ακόμα περισσότερο οι σχέσεις μας. Και τώρα έχουμε την εξής κατάσταση. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση Είμαστε πολύ δραστήριοι στην περιοχή γύρω από την Ταϊβάν, εμπορικό πώ. Εδώ και λίγου μήνε έχουμε τη ε, Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών με την Νότιο Κορέα. Έχουμε αρχίσει διαπραγματεύσει για Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με την Ιαπωνία. Έχουμε εμπορικέ σχέσεις με την Κίνα, τώρα μόλις το συζητούσαμε, και θα συνάψουμε και θα ε, εντείνουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μας με την υπηρετική Κίνα. Γενικά στην Ασία δραστηριοποιούμαστε, έχουμε διαπραγματεύσεις και με πολλές άλλες χώρες. Από την άλλη όμως μέχρι τώρα δεν βρήκαμε δυνατότητα να συσφίξουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με την Ταϊβάν. Και τώρα δεν έχει νόημα σίγουρα να μιλάμε για συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ούτε κατά διάνοια με την Ταϊβάν, αλλά από κοινού να προβληματιστούμε. Έχουμε καλές εμπορικέ σχέσεις με την Ταϊβάν, πώ θα τι καλλιεργήσουμε, θα τι διευρύνουμε και πώ θα αποφύγουμε σε αυτό το περιβάλλον που σας περιέγραψα, δηλαδή που έχουμε με πολλές γειτονικές χώρες και όμορες, άμεσες, ε, σύσφυξη των εμπορικών σχέσεων και έχουν και παράγουν τα ίδια βιομηχανικά προϊόντα. Και οι δικές μας εταιρείε στην Ταϊβάν είναι πάρα πολύ δραστήριες και ενεργές. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνει και οι Ευρωπαίοι επενδυτές είναι από τους μεγαλύτερους στην Ταϊβάν. Θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Τι θα κάνουμε και πώς θα εντείνουμε και θα συσφίξουμε τις εμπορικές μας σχέσεις. Γι' αυτό ερωτούμε σήμερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πώ εκτιμά τι εμπορικέ μα σχέσει με την Ταϊβάν τι δυνατότητες βλέπει να συσφίξουμε τις σχέσεις αυτές, να τις βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω, ε, δεδομένης και της κατάστασης που σας περιέγραψα και των προσεχών διαπραγματεύσεων με την Κίνα και τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε να μην απομονωθεί σε αυτό το τρίγωνο ή το πολύγωνο των διαφόρων εμπορικών μας σχέσεων που έχουμε με τις διαφόρες χώρες. Γι' αυτό ακριβώς μετά τη συζήτηση με την Κίνα, για την Κίνα, ε, χαίρομαι πάρα πολύ που συζητούμε αυτή την ερώτηση και ευχαριστώ ε, όλες τις πολιτικές ομάδες που συμφωνήσαμε για αυτή τη σειρά στη διάταξη των εργασιών να ε, ανταλλάξουμε απόψεις ε, ειλικρινά και ε, να δούμε πώς θα συνεχίσουμε τις σχέση μας με την Ταϊβάν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Επίτροπος έχει το λόγο. Κύριε Ντεχέχτη, παρακαλώ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κασπάρη, αξιότιμοι κύριοι ευρωβουλευτέ μολι πριν δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε, απάντησε μάλλον, σε μια προφορική ερώτηση για τι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ταϊβάν. Πολλά από αυτά που υπόθηκαν τότε εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα. Ωστόσο, η Ταϊβάν έχει ανέβει Συγγνώμη, έχει κατέβει από τη 15η θέση στην 23η θέση ως εμπορικός εταίρος ε, της Ένωσης. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, παραμένει ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Ταϊβάν. Αν δείτε τα στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, οι σχέσεις οι εμπορικές μεταξύ Ένωσης και Ταϊβάν έχει ακολουθήσει ανωδική τάση, όπως αυτή τον ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Παρά την πρόσφατη παρακμή που οφείλεται στην οικονομική κρίση του 2008, και μετέπειτα. Έχουμε ολοκληρωμένο διάλογο. Οι ανώτατοι υπάλληλοι συναντώνται τουλάχιστον μια φορά ετησίω και μιλούν για διάφορα θέματα, τεχνικού φραγμούς στο εμπόριο, ε, δικαιώματα πραγματικά, γεωγραφικές, ε, ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης, δημόσιες προμήθειες, ε, φαρμακευτικά θέματα. Ο διάλογός μας εστιάζει περισσότερο τους μη ε, δοσμολογικούς φραγμούς και δίνει αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές. Αμοιβαία κατανόηση που οικοδομείται σε αυτές τις συνεδριάσεις και η συζήτηση θεμάτων που διαφορετικά θα αποτελούσαν φραγμό για, τον, για το εμπόριο έχουν οδηγήσει στη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος που προστατεύει την, την πνευματική ιδιοκτησία και που οδηγεί σε αμοιβαίες επενδυτικές ροές. Η Επιτροπή έχει επαφές, ε, διαπραγματεύσεις με την Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και την Ιαπωνία. Και επιπλέον αρχίζουμε επενδυτικές διαπραγματεύσεις με την ε, υπηρετική Κίνα, πράγμα που μόλις συζητήσαμε εδώ στην Ολομέλεια. Πρέπει να εστιάσουμε στην ε, ατζέντα μας. Αργότερα θα χρειαστεί να αξιολογήσουμε διάφορους τρόπους για να ε, ε, ενισχύσουμε το εμπόριο με την Ταϊβάν μέσω επενδυτικών συμφωνιών, που θα καλύπτουν την πρόσβαση στην αγορά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέφτ. Τώρα οι μιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, ο κύριος Στάσνη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η έγκριση του ψηφίσματος για να ανοίξουμε εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ταϊβάν είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για να ενισχύσουμε τις σχέσεις ε, οικονομικά και πολιτιστικά. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες ε, το διμερές εμπόριο ε, έχει πολλαπλασιαστεί επί τέσσερα και είναι περίπου 40 δισεκατομμύρια το 2011. Ακόμα και με τον τρόπο αυτό το εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Ταϊουάν είναι πολύ κάτω από τις δυνατότητες του. Ε, το, η Ταϊουάν είναι μια εύρωστη, μια στερεή ε, δημοκρατία και μια εύρωστη οικονομία. Ε, στην Επιτροπή Ίντα είμαστε υπέρ μια χειρότερε εμπορικής συμφωνίε ε, για να συλλέξουμε ωφέλη. Δεν θέλουμε ε, να είμαστε οι πρώτοι. Το μήνυμα είναι σαφές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε να προκαλέσει την Κίνα και δεν θέλει ε, να πειράξει με την Ταϊουάν άλλες χώρες με τη, με Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών, Κορέα, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη διαπραγματεύονται ή έχουν συνάψει επενδύσεις ε, με την και εμπορικές συμφωνίες ε, με την Ταϊουάν. Μπορεί η Ευρώπη να μείνει πίσω. Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση είναι σαφής. Για να ωφεληθούν οι πολίτες από τις δύο πλευρές οι για στενότερη και βαθύτερη ε, συμφωνία μεταξύ Ευρώπης και Ταϊουάν θα πρέπει να αρχίσουν πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στάσνη. Ο συνάδελφος Μορέιρα, για ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ταϊβάν ε, έχουν ακόμα πολύ χώρο να αναπτυχθούν. Παρότι αναπτύσσονται διαρκώς και ε, πολλαπλασιάστηκαν επί 12 την τελευταία 20 ετία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ της ευάθεσης των σχέσεων αυτών. Το ψήφισμα της, ε, της Επιτροπής ε, Διεθνούς Εμπορίου τονίζει ιδιαίτερα τη δυνατότητα διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας επενδυτικής συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, γίνονται διαπραγματεύσει με την Κίνα και δεν υπάρχει λόγος για να μην γίνει μια άλλη τέτοια συμφωνία με την Ταϊβάν από τη στιγμή που θα πληρούνται οι προποθέσει. Τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να, να συνάψει επενδυτικές συμφωνίες αμοιβαία απελευθέρωση επενδύσεων, δηλαδή πρόσβαση στην αγορά και προστασία των επενδυτών. Αν και δεν εντάσσεται στου καθορισμένου προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο 2010 στην ανακοίνωση ε, για τι επενδύσει, δεν υπάρχει κανένα λόγο ε, για να εξαιρείται η Ταϊβάν από την ατζέντα τη ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Μαρέρα. Και τώρα ο κύριος Κασάκ για δύο λεπτά господин председател уважаеми господин комисар аз Αξιότιμε κύριε Επίτροπε, εγώ δεν θέλω να επαναλάβω όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις εμπορικές μας σχέσεις με την Ταϊβάν. Είναι σαφές ότι είμαστε πίσω από το πραγματικό δυναμικό των οικονομικών μας σχέσεων. Χρειάζεται να τις εμβαθύνουμε και να ε, επενδύσουμε στις ε, ήδη καλές ε, οικονομικές σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στους δύο εταίρους, ώστε να αναπτυχθεί η βιομηχανία, η τεχνολογία της πληροφορικής, καθώς και η τεχνολογία της πράσινης ενέργειας. Θα δοθούν έτσι ευκαιρίες για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας που προσφέρουν ανάπτυξη και για τους δύο εταίρους Ταυτόχρονα θα ήθελα να πω ότι η οικοδομητική προσέγγιση της Ταϊβάν οδήγησε στην υπογραφή 31 δημερών συμφωνιών συμπεριλαμβανομένης της Κίνας και της Ιαπωνίας. Όλα αυτά αποδεικνύουν πως η Ταϊβάν είναι έτοιμη να συνάψει παρόμοιες συμφωνίες με άλλους εταίρους συμφωνίες που βασίζονται στο πολυμερές εμπορικό σύστημα του ΠΟΕ. Είμαι πεπισμένος ότι οι μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες ανάμεσα στην Ένωση και την Ταϊβάν θα αυξήσουν τις εξαγωγές της Ένωσης κατά 12 δις ετησίως. Γι' αυτό κάνω έκκληση προς την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία και να βρει τη βάση για τη διαπραγμάτευση μιας δημερούσης συμφωνίας. Η Κομισιόν δεν θα πρέπει να υποτιμά τα αμοιβαία ωφέλη μιας τέτοιας συμφωνίας με την Ένωση. Είμαι πεπισμένος πως η Ταϊβάν θα πρέπει να μείνει πίσω σε σύγκριση με την Κίνα. Γιατί μια συμφωνία τέτοιου τύπου στηρίζει τη δημοκρατία και το κοινωνικό πλουραλισμό σε μια χώρα όπως η Ταϊβάν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καζάκ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Ε, Εμεί οι πράσινοι δεν συμμεριζόμαστε αυτή τη βιασύνη τώρα να ε, ε, κάνουμε συμφωνία με την Ταϊβάν. Ήδη υπάρχουν επενδύσεις εκεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα είναι ο πρώτος επενδυτής, ξένος και οι δύο οικονομίες είναι πολύ καλά ολοκληρωμένε, οπότε δεν πρέπει επιγόντως να κάνουμε κάτι. Επανειλημμένα ως Κοινοβούλιο δηλώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου θα πρέπει να θέτει προτεραιότητες στις διαπραγματεύσεις τις εμπορικές. Ακριβώς γιατί έχουν και περιορισμένο προσωπικό. Έχουμε διαπραγματεύσει με Ηνωμένε Πολιτείε, Καναδά, Ινδία, για να σα πω μερικέ μόνο χώρε. Ω κοινοβούλιο στριμωχνόμαστε επιπλέον όταν πρέπει να τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε να αναλύουμε και να παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις. Και έχουμε και την αξίωση να παρακολουθούμε και μετά τη σύναψη συμφωνίας, αυτές τις συμφωνίες. Και εμείς οι πράσινοι θεωρούμε ότι είναι καλό βέβαια να μην ξεχνούμε τις σχέσεις μας με την Ταϊβάν Ιδιαίτερα όταν διαπραγματευόμαστε εμπορική συμφωνία και επενδυτική με την Κίνα. Καλά κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καλωσορίζει και να χαιρετίζει τι θετικέ εξελίξει ε, στην Ταϊφάν για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου και να το διατρανώνει κιόλα. Για μα είναι σημαντικό οι διμερεί σχέσει να υποστηρίζονται και από αυτό το πρίσμα και όχι μόνο από το οικονομικό. Λοιπόν, εφόσον επιθυμούμε ενισχυμένο διάλογο, να μην είναι μόνο για εμπορικά θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλα. Για δύο λεπτά ο κύριος Στάνο. Κύριε Πρόεδρε, ως πρόεδρος της ομάδας φιλίας με την Ταϊουάν. Εδώ και χρόνια κάλεσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση να απαντήσουμε, να αντιδράσουμε στο δυναμισμό της Ταϊουάν και μια τέτοια συμφωνία θα έχει μεγάλο όφελος και για τους δύο. Είναι ένα από τα οικονομικά θαύματα του 20ου αιώνα μετά από την απικιακή εποχή έχει γίνει μια κινητήριος δύναμη και παράγει πάρα πολλά από τα αγαθά που καταναλώνεται σήμερα. Έχετε ουίσκι, έχετε ρούχα από την χώρα αυτή. Η βελτίωση των εμπορικών σχέσεων με την Ταϊουάν έχει νόημα και για αυτούς και για μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων είναι μεγάλο επίτευγμα αν θεωρήσουμε τον ανταγωνισμό σε αυτήν την Ήπειρο και τον μικρό πληθυσμό της Ταϊουάν σε σχέση με τον πληθυσμό της Κίνας 58 φορές μεγαλύτερος ο πληθυσμός αλλά το εμπόριο 11 φορές μεγαλύτερο. θα πρέπει να συγχαρούμε τον Πρόεδρο για τον διάλογο με το Πεκίνο που έκανε τόσα πολλά ε, για να προωθήσει το εμπόριο με την Κίνα. Είχε φέτος ε, μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών με την ε, Νέα Ζηλανδία και μια χώρα που δεν την αναγνωρίζει. Έχουμε μια δημοκρατία εύρωστη που δεν θα πρέπει να είναι όμοιρος των, της καταστάσεως θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την Ταϊουάν να συμμετάσχει στον ΙΚΑΟ, στον ΠΟΕ και πρέπει να χαιρετήσουμε ε, την, ε, την εταιρική σχέση ε, που βασίζεται στην δημοκρατία και στην υπεροχή του δικαίου. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Επιτρέπετε ερώτηση με για κάρτα από τον κύριο Σόλτς. question of colleague Έχει να σας ρωτήσει ο κύριος Σόλτς. Θέλετε να δεχτείτε το ερώτημά του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφε Τάνοκ, ε, πώς αξιολογείτε την πολιτική της μίας Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι διπλά κοινική ε, η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από αρχές της δεκαετίας του 90 ε, ε, επενδυτές από τη Ταϊβάν παίρνουν μεγάλο τμήμα της πίτας της κινέζικης ανάπτυξης και με μεγάλα κέρδη. Και υπάρχει και μια εταιρεία που λέγεται Foxconn που είναι ε, της Ταϊβάν και έχει κακές εμπορικές και κοινωνικές συνθήκες. Μα δεν ακούσατε τι σα είπα. Εγώ για τη Νέα Ζηλανδία είπα ότι μιλάει για την πολιτική τη μία Κίνα. δεν αναγνωρίζει την Ταϊβάν ω ανεξάρτητο κράτο. αλλά με το έδαφο τη Ταϊβάν έχει συμφωνία εμπορική και ανήκει και η Ταϊβάν στον ΠΟΕ. Οι περισσότερε χώρε που δεν την έχουν αναγνωρίσει ω ανεξάρτητη συνεργάζονται. Ζούμε σε έναν κόσμο επικοδομητική αμφισημία ω προ την Ταϊβάν. Έχουμε κοινέ αξίε και είτε το, την αναγνωρίζει κανεί είτε όχι, που 30 χώρε την έχουν αναγνωρίσει, δεν έχει σημασία. Αυτό που θέλουμε εμεί καλύτερε εμπορικέ σχέσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ και τώρα ο συνάδελφο Μπέλτερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ω Ολλανδό, έχω επίγνωση του γεγονότο ότι συνδεόμαστε ιστορικά με την Ταϊβάν, Φορμόζα. Από το 1624 ε, συνδεόμαστε. Έχουμε τεράστιες σχέσεις και προαιώνιες. Ε, πριν από δύο χρόνια εδώ στην Ολομέλεια, το είπε και ο Επίτροπος, έγινε συζήτηση για τις εμπορικές σχέσεις με την Ταϊβάν. Και τότε ζήτησα αναβάθμιση των σχέσεων μας, των εμπορικών ή ε, μέτρα προώθησης του εμπορίου. Τώρα, δύο χρόνια αργότερα, δυστυχώς έρχομαι να διαπιστώσω ότι έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Και ούτε εμπορικά πλεονεκτήματα έχουμε, Τώρα ε, ε, ακολουθούμε την ε, πορεία Πεκίνου Ταϊπέη και προσπαθούμε να βαθμίσουμε τις σχέσεις μας, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε τουλάχιστον δύο χρόνια αργότερα. Ευχαριστώ για μισή λεπτό. Τελευταίος εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων, ο Γονής. Ε, Αγαπητέ συνάδελφε Μπέλτερ, οι Πορτογάλοι συναδέλφοι, συνάδελφοι θα σας πούνε ότι είχαν τις πρώτες σχέσεις με την Ταϊουάν, τις πιο παλιές, διότι φτάσανε πριν από τους Ολλανδούς. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό σήμερα. Η Ταϊουάν ευτυχώς ε, ξέφυγε από τον κομμουνισμό το 1949 και συνεπώς ε, με την ευφυΐα του πληθυσμού, την πειθαρχία, τις παραδοσιακές αξίες, την καλλιέργεια των ατόμων γνώρισε ταχύτατη ανάπτυξη που θα μπορούσε να είναι αυτή της Κίνας αν δεν υπήρχε ο μαοϊσμός. Το επίπεδο ζωής στην Ταϊουάν αυξήθηκε πάρα πολύ και ο ανταγωνισμός με την Ταϊουάν, ο ανταγωνισμός που είναι ε, το απαραίτητο αντίβαρο ε, στις ε, διεθνείς σχέσεις δεν βασίζεται στο κοινωνικό dumping όπως συμβαίνει με άλλες χώρες όπως με την μεγάλη κομμουνιστική χώρα την Κίνα την υπηρετική που έγινε παράδεισος του άγριου καπιταλισμού. Βεβαίως τα, οι ελεύθερες συναλλαγές έχουν ωφέλη, πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν πρέπει να διστάζουμε να έχουμε επίσημες σχέσεις με την Ταϊουάν, να θέσουμε τέρμα στην υποκρισία και να αφήσουμε τους λαούς των δύο χωρών να αποφασίσουν μόνοι τους για μια επανόνηση μιας ε, Κίνας ελεύθερης ε, ή μιας ανεξαρτησίας. Πρέπει να υποστηρίξουμε την υποψηφιότητα της Ταϊουάν στα όργανα και στους οργανισμούς Οργανισμούς των Ηνωμένων τους ε, υπόλοιπους εγγεγραμμένους ομιλητές και θα δώσω πρώτα το λόγο στη συνάδελφο Άντρη Κένε για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Έχουμε βεβαίως βάσεις και οι ευρωπαϊκές εταιρείες ασχολούνται με πολλούς τομείς της οικονομίας Πάρα πολλές εταιρείες έχουν κοινέ επιχειρήσεις, joint ventures, οι Ευρωπαίοι έχουν περίπου επενδύσει 30 δισεκατομμύρια στην ε, Ταϊουάν ε, και η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη ομάδα ε, ξένων επενδυτών. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ταϊουάν έχουν επίσης συνεργασία με την υπηρετική Κίνα για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα. Θα ήθελα τώρα να στραφώ σε μερικές πολιτικές απόψεις της συζήτηση. Ξέρουμε πόσο η διεθνής κατάσταση της Ταϊουάν είναι περίπλοκη και αυτό επηρεάζει τις εμπορικές της σχέσεις. Είναι μια ειρηνική χώρα, δημοκρατική, πρέπει λοιπόν να αποτελέσει όλο και περισσότερο μέρος της παγκοσμιοποίησης και η ένταξη στην παγκόσμια οικονομία είναι ε, η συμφωνία με την Κίνα, η ΕΠΦΑ, η οποία αποδεικνύει ότι η ε, Κίνα de facto την έχει περιλάβει στο διεθνές εμπόριο και έχει αναγνωρίσει την οικονομική της ανάπτυξη εν κατακλείδη η θέση της στην παγκόσμια οικονομία απαιτεί στενότερη σχέση με την Ευρώπη. Η συμφωνία έχει σαφή στόχο. Η ΕΠΦΑ, η Ουκορία ε, και η ζώνη ελευθέρων συναλλαγών με τη Σιγκαπούρη δείχνει ότι ήρθε η στιγμή να έχουμε μια συμφωνία με την Ταϊουάν και η Ταϊουάν και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αφεληθούν από μια εμπορική συμφωνία όχι μόνο για την αύξηση του εμπορίου αλλά ε, για την συμμετοχή αυτή στο τρίγωνο σχέσεων με την Κίνα επίσης. Ε, Μετά από την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα και στην Κίνα που μόλις συζητήσαμε, πιστεύω ότι είναι και ώρα, είναι απαραίτητο να προβούμε σε μια επιλογή και να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με την Ταϊβάν. Οι όγκοι τάσεις έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αν και είναι κάτω από το πραγματικό δυναμικό. Η Ένωση επενδύει πολύ στην Ταϊβάν, είναι μάλιστα ανάμεσα στους βασικούς ξένους επενδυτές. Οι επιχειρήσεις μας ήδη εδώ και καιρό έχουν προβεί σε εμπορικέ συμφωνίε ε, με βάση την πραγματικότητα τη Ταϊβάν. Αλλά λείπει ε, το θεσμικό πλαίσιο και οι πολιτικοί και οι θεσμοί μπορεί να φτάσουν πολύ αργά σε σχέση με τα οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα τα οποία προχωρούν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να οθήσουμε έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να δουλέψει για μια εμπορική επενδυτική συμφωνία με την Ταϊβάν, να ξεπεράσουμε του δισταγμούς και να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα Φαίνεται να είναι και μια ευκαιρία για να φτιάξουμε την πολιτική, την εξωτερική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα λοιπά. Η Ταβάν είναι μια εκπληκτική πραγματικότητα όσον αφορά τη δημοκρατική διαδικασία αλλά και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και αξίζει μια νέα προσοχή από πλευρά της Ένωσης. Πιστεύω λοιπόν πως θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η δουλειά που μπορεί να αναλάβει η Κομισιόν υπό το φως και των νέων ε, ε, παφών που έχουμε με την Κίνα για να ξεκινήσουμε ξεκινήσει και με το Ταϊβάν. Ε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οικονομικέ και εμπορικέ συμφωνίες που έχουν ξεκινήσει με διμερεί συμφωνίες ε, ήδη υπογεγραμμένε ε, με πολλές χώρες όπως και με την ε, λαϊκή δημοκρατία της Κίνα, Αλλά η Ταϊβάν είναι και μια δημοκρατική χώρα. Μιλάμε την ίδια γλώσσα για μια πλουραλιστική συμμετοχική κουλτούρα. Ε, μιλάμε για διμερή συμφωνία επενδυτική με το Πεκίνο. Είναι αδύνατο να αφήσουμε πίσω ένα σαφές και φιλόδοξο ρυθμιστικό πλαίσιο ανάμεσα στην Ένωση και την ΤΑΙΠΕ. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό. Υπάρχουν ε, τα νούμερα των ανταλλαγών, ε, ποιοτικά προϊόντα. Η Ταϊβάν είναι μια από τις χώρες με τα μεγαλύτερες ευρεσιτεχνίες κατά κεφαλήν. Ε, δεύτερον, οι αξίε μα το να έχουμε εμπόριο με μια δημοκρατία είναι πάντοτε πιο πλεονεκτικό και από ηθική άποψη από ότι να το κάνουμε αισθάνομαι με μια χώρα που ακόμα γνωρίζει την ε, κουλτούρα του ενός και μόνου κόμματο. Εξάλλου είναι και θέμα πολιτική. Η Ταϊβάν υπάρχει ως κράτος. Υπάρχει, δεν αναγνωρίζεται από την Ένωση, αλλά υπάρχει και είναι ανεξάρτητο εδώ και χρόνια. Το να εμποδίζεται η πρόσβαση στι διεθνούς οργανισμούς όπως ε, με τον, προ... τον Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας ε, πρόσφατα είναι και αυτό ο καρπός μιας πολιτικής και των σχέσεων δυνάμεων στην περιοχή. Αλλά δεν είναι η πραγματικότητα αυτή της Ταϊβάν και έπειτα εδώ μιλάμε για αγορές πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταϊβάν έχει μεγάλη σημασία. Οι εμπορικές μας συναλλαγές τα τελευταία 20 χρόνια είχαν εντυπωσιακή αύξηση και χαίρομαι γιατί η Ταϊβάν καταλαμβάνει μια ιδιαίτερη θέση και δεν είναι εύκολη θέση της διεθνώς γιατί πιέζει συνεχώς η λεγόμενη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας. Σε ε, αντίθεση με την λαϊκή λεγόμενη ε, δημοκρατία, η Ταϊβάν είναι δημοκρατία ουσιαστική και πρέπει να το τονίζουμε συνεχώς. Και ως Ευρωπαϊκή Ένωση καλό θα είναι να αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε για μια τέτοια συμφωνία. Θα είναι εποφελής και θα έχει μεγάλα πλεονεκτήματα και για τις δύο πλευρές και θα μπορέσει να βγει από τη διπλωματική απομόνωση η Ταϊβάν. Και αυτά θα πρέπει να τα καταλάβει σαφέστατα η κομμουνιστική Κίνα. Το πλεονέκτημα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες θα είναι καλύτερη πρόσβαση στις αγορές της Ταϊβάν και αυτό θα είναι μια αρχή για καλύτερη προστασία ε, της πνευματικής ιδιοκτησίας των ευρωπαϊκών εταιριών. Γιατί μπορεί να έχουν λάβει μέτρα οι αρχές στην Ταϊβάν, απομένει πολύς δρόμος ακόμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Συνάδελφος Λίζεκ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Όπως γνωρίζουν πολλοί από σας παρόντες εδώ στην αίθουσα, είχα και εγώ την ευκαιρία να επισκεφτώ την Ταϊβάν, μαζί σα άλλωστε. Και τι είδα εκεί πριν από μήνε. Κυρίως ότι είναι μια χώρα δημοκρατική. Είδα εκπροσώπους των δύο μεγάλων πολιτικών κομμάτων και μάλιστα αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει ότι είναι μια κανονική δημοκρατία με κανονικό πολιτικό παιχνίδι και κανονικές εκλογές. Αυτό θα πρέπει να το τονίζουμε γιατί δεν ισχύει παντού στις ασιατικές χώρες αυτό. Ε, δεν επικρατούν παντού τέτοιες συνθήκες δημοκρατίας. Επίσης, είδα πάρα πολύ προηγμένη τεχνολογία, πολύ ανεπτυγμένη οικονομία και πολλοί από εσά επίσης σήμερα μίλησαν για τη σχέση μας με την Κίνα. Εδώ θα πρέπει να γνωρίζουμε μερικές πραγματικότητες των περασμένων μηνών και να μας απασχολούν σήμερα και κάθε μέρα προσγειώνονται δεκάδες αεροπλάνων από την Κίνα στην Ταϊβάν και το αντίστροφο από την Ταϊπέη στην Κίνα, στο Πεκίνο και στη Σανγκάη. Ε, δεκάδες χιλιάδες είναι Κινέζοι επισκέπτες και τουρίστες στην Ταϊβάν και ε, δισεκατομμύρια δολαρίων ε, επενδύουν Ταϊβανέζοι πλέον στη λαϊκή δημοκρατία. Και όταν λέμε ότι η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας είναι ο παριθμόν ένα εξαγωγέας, θα πρέπει να κοιτάξουμε τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες που εξάγουν και σε αυτό το κατάλογο οι 7 από τις 10 και οι πρώτες 5 είναι εταιρείε από την Ταϊβάν παρακαλώ που έχουν μεταφέρει την τεχνολογία τους και έχουν επενδύσει τα χρήματά τους στη λαϊκή δημοκρατία. Όλα θα, θα πρέπει να τα γνωρίζουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συσφίξει τη σχέση της με την Ταϊβάν χωρίς καμιά αμφιβολία. Ευχαριστώ. Λίζε, η συνάδελφος Μαρία Μπαντία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε. εν ώψη ε, της σύσφυξη των εμπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταϊβάν τις τελευταίες δεκαετίες, ε, πρέπει σήμερα να ανταποκριθεί θετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση στη βούληση που έχει εκφράσει η Ταϊβάν ε, για μελλοντική συμφωνία. Έτσι θα εδρεωθούν και οι δημοκρατικές δομές στη χώρα όπως έχει γίνει με την Νότιο Κορέα και με άλλες χώρες της περιοχής. Και έτσι θα εμβαθύνουμε και την ε, αμοιβαία υποφελή σχέση μα και για τι δύο οικονομίε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προστασία των επενδύσεων και την πρόσβαση στην αγορά. Υπό την έννοια αυτή, μεγαλύτερη όθηση και προώθηση ε, των τεχνολογιών ε, θα σημάνει βελτίωση για τις οικονομίες. Βέβαια θα πρέπει να γίνεται πάντα με ε, τους κανόνες της αμοιβαιότητας του πολυμερούς εμπορίου ε, με κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρε και κοινωνική εταιρική ευθύνη. Ευχαριστώ. Το πολύ, ο συνάδελφος Γκραχαμ Γουότσον. Πρόεδρε, η τελευταία μας συζήτηση αφορούσε την πρώτη αυτόνομη επενδυτική συμφωνία Τη Ένωση από τότε που τη δόθηκε αρμοδιότητα από την συνθήκη τη Λισαβόνα. Δεν θα είναι ιστορική στιγμή. Δεν πρέπει να την αφήσουμε μόνη και έρημη αυτή την πρώτη ε, συμφωνία. Το νησί αυτό είναι γνωστό στους Ευρωπαίους επιχειρηματίες. Έχουμε εμπορευτεί ε, για χρόνια και γιατί. Αυτό το ο ασιατικός είναι ένα λιοντάρι της ελεύθερης αγοράς. Έχουμε τακτικούς διαλόγους για τις επενδύσεις και το εμπόριο, αλλά οι διμερείς εμπορικοί όγκοι υπολείπονται. Ε, και το δυναμικό για διμερείς επενδύσεις είναι τεράστιο. Ε, Εμεί ε, μιλάμε για αξίε και για μια συμφωνία με τη λαϊκή δημοκρατία τη Κίνα. Ε, η συνθήκη μα δίνει τη δυνατότητα να στηρίξουμε τη δημοκρατική Ταϊβάν. Και αν αποφασίσουμε συμφωνία με την Κίνα ω δρόμο για να αυξήσουμε τι επενδύσει και τα εμπορικά ισοζύγια, τον ίδιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε και για την Ταϊβάν και να επιτρέψουμε και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επενδύσει εκεί. Ε, καλό λοιπόν να, την Κομισιόν να προτείνει μια παράλληλη win-win ε, κατάσταση για τους, τα δύο μέρη, παράλληλη συμφωνία με την Ταϊβάν και για τους επενδυτές και για την αύξηση του όγκου και της ποιότητας των επενδυτικών ροών. Σα ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Γουότσο. Να υπάρχει μπλε κάρτα από τον συνάδελφο Καζάκ. Τη δέχεστε? Ο κύριος Καζάκ λοιπόν. Sir Graham Watson, като Επειδή είστε κάποιο που γνωρίζετε πολύ καλά την Κίνα, αναφέρατε πόσο σημαντικό είναι να αναβαθμιστούν οι σχέσει μα με την Ταϊβάν στο τομέα του εμπορίου. Ε, αλλά ξέρετε πόσο λεπτή είναι η κατάσταση με την ε, Ταϊβάν σε σχέση με την ε, Κίνα. Τι Ποια νομίζετε ότι θα είναι η ανταπόκριση της Κίνας αν η Ευρωπαϊκή Ένωση λάβει απόφαση και βελτίωση των εμπορικών σχέσεων με την Ταϊβάν. Θα πρέπει να φοβόμαστε, φοβόμαστε την αντίδραση της Κίνας. Πρόεδρε, νομίζω πως ο εξαιρετικός φίλος κ. Καζάκ άγγιξε κάτι που σίγουρα θα είναι ένας φόβος στο μυαλό κάποιων από τους ηγέτες των κρατών μελών αλλά η Ένωση θα πρέπει να δείξει τόλμη σε αυτά τα θέματα. Η Κίνα επισήμω δεν έχει αντίρρηση στο εμπόριο με την Ταϊβάν, οπότε δεν μπορεί να έχει ρεαλιστικέ ή ε, αντιρρήσει για αυτή ε, τη συμφωνία με την Ταϊβάν. Είναι προ το δικό μα συμφέρον να οθήσουμε ε, τι αξίε μα και άρα εμπόριο με όλε τι χώρε και να, να αναγνωρίσουμε ότι με τι δημοκρατίε έχουμε πολλά πιο πολλά κοινά από ότι με αυτέ τι χώρε που δεν είναι δημοκρατικέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε με, για μια συμφωνία με τη Σιγκαπούρη, την Κορέα και θα διαπραγματευτούμε με την Κίνα. Θα έχουμε λοιπόν φθηνότερα αγαθά για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταϊουάν, μια σύγχρονη δημοκρατία, έβδομος μεγαλύτερος εταίρος και δεν έχουμε εμπορική συμφωνία. Γιατί νομίζω λόγω φόβου. Φοβούμεθα την αντίδραση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, διότι για το Πεκίνο δεν υπάρχει η Ταϊουάν. Είναι μια επαρχία και λόγω αυτού ε, νομίζω ότι ε, έχει, βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Η Νέα Ζηλανδία σύναψε συμφωνία, έχουμε άλλες συμφωνίες επενδύσεων και αν θέλουμε να βασιστούμε στην Ταϊουάν, να έχουμε εμπιστοσύνη στην Ταϊουάν, ε, δεν ε, θα διακινδύνευαν να διαπραγματευτούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν αυτό, με αυτό διακινδύνευαν τις σχέσεις με την Κίνα εφόσον έχουμε και συμφωνία με το μεγαλύτερο ανταγωνιστή τους. Γιατί όχι, η Ταϊουάν κάνει το ίδιο με τους ανταγωνιστές, αλλά τώρα έχει πρόσβαση στην Ευρώπη. Δεν πρέπει να την παρεμποδίσουμε να έχει πρόσβαση στην μεγαλύτερη αγορά επειδή σεβόμεθα μια μεγάλη δικτατορία γειτονική αντί να σεβόμεθα την μικρή δημοκρατία. Έχουμε τα θέματα εδώ τα οποία είναι ηθικής φύσεως για το καλό της Ταϊουάν και το δικό μας θα πρέπει να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις για φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες και το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ο δικός μας φόβος για το τι θα συμβεί. Ναι, θα αυξήσουμε τις σχέσεις μας με την Ασιατική Ήπειρο με διαπραγματεύσεις φιλόδοξων εμπορικών συμφωνιών. Πολλές γειτονικές χώρες ε, της Ταϊουάν, η Ταϊλάνδη, η Κορέα έχουν ε, ε, προοπτικές που υπόσχονται πολλά για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να απομονώσουμε αυτήν ε, την χώρα και να την αποκλείσουμε από οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να, να διαπραγματευτεί με βάση τους διεθνείς κανόνες. Οι διεθνείς κανόνες επιτρέπουν στην ε, Ταϊουάν επικοδομητική πολιτική. Έχουν 19 συμφωνίες με την Κίνα και 31 συμφωνίες με άλλες χώρες. Αυτό είναι, είναι μέρος ε, του ε, ΠΟΕ και του Ασιατικού Φόρουμ. Λοιπόν, υποστηρίζω τη διεύρυνση των ε, σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ταϊουάν. Ευχαριστώ κύριε Τζεζέμερα. Είναι η 18η εμπορική δύναμη στον κόσμο η Ταϊβάν. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταϊβάν συνεπώς είναι πάρα πολύ σημαντικέ και απαραίτητε. Πάνω από 12 φορές ε, αυξήθηκε ε, τις τελευταίες δεκαετίες το εμπόριο. Και τώρα έχουμε τη δυνατότητα με μια συμφωνία να ευρεώσουμε και να ενισχύσουμε τις σχέσεις αυτές οικονομικοί παράγοντες, κυρίες και κύριοι, μαζί με τις υψηλές προδιαγραφές δημοκρατίας καθιστούν την Ταϊβάν πολύ σημαντικό στρατηγικό εταίρο. Γι' αυτό θα ήθελα να παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Ντεχόχτ να αρχίσουν ε, διαπραγματεύσεις εμπορίου και επενδύσεων με την Ταϊβάν. Να σας δώσω μερικά αριθμητικά στοιχεία για να το τονίσω αυτό. Το 2002 ε, μπήκε πλήρως στον ΠΟΕ το 2010 εδώ στο Κοινοβούλιο εγκρίθηκε η απελευθέρωση των θεωρήσεων διαβατήριο και μου και εισηγητής. Τον Ιούνιο του 2010 υπέγραψε με τη Λαϊκή Δημοκρατία η Ταϊβάν μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών και ε, σχετικά με την πνευματική διοκτησία. Επιπλέον, έχει 31 διμερείς επενδυτικές συμφωνίες με πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένες της Ιαπωνίας. Ε, ξανάρχισε τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείε. και ε, ε, με ε, άλλες χώρες του κόσμου μπορεί να μην έχουν με τη Νέα Ζηλανδία διπλωματικές σχέσεις αλλά έχουν συνάψει εμπορική συμφωνία. Τέλος κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, η Ταϊβάν έχει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών με τον Παναμά, το Σαλβαδόρ, Ονδούρα, Γουατεμάλα, και Νικαράγουα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει το συντομότερο τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Επενδύσεων και Εμπορίου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, I think that colleague... Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο συνάδελφος Λούχαν είναι απόν, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στη διαδικασία κατσιά και όταν έρθει ο κύριος Λούχαν μπορεί αργότερα να του δοθεί ο λόγος. Πρώτα απ' όλα το λόγο στον συνάδελφο Κέλλη. uachtaráin arís agus is bheith ar an ábhar seo chomh maith. I think. Uh, Ο πολύ έμπειρος κ. Στάνοκ τα όλα όταν μίλησε για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ταϊβάν. Αναφέρθηκε στον οικονομικό της δυναμισμό, το οικονομικό θαύμα της Ταϊβάν και την βελτίωση βελτίωση ε, και μάλλον και ε, ότι έχει απόλυτο νόημα αυτή η εμπορική συμφωνία. Και ναι, θα πρέπει ταυτόχρονα με την Κίνα να συζητήσουμε. Δεν αποκλείει μία την άλλη και είναι σωστό να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις και με τις δύο ειδικά όσον αφορά το εμπόριο. Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη το γεγονός ότι η δημοκρατική, ε, ε, ότι η Ταϊβάν είναι δημοκρατική χώρα όπως και εμείς και πρέπει να τους βοηθήσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό και ε, είναι πρόσδεκτες οι απόψινές συζητήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μορβά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Αν πάτε σε Βουδαπέστη περίπατο ή επισκεφτείτε μια άλλη ουγγρική πόλη, θα δείτε σίγουρα κάτι πάρα πολύ ε, θλιβερό. Υπάρχουν ε, πολύ μικρομεσαίοι ε, που έχουν βάλει λουκέτο. Υπάρχουν δάσκαλοι και ε, φτωχοί άνθρωποι που βλέπουν τη ζωή τους να καταστρέφεται ή να απειλείται. Για ποιο λόγο? δεν μπόρεσαν να αντέξουν τον ανταγωνισμό. απέναντι σε μεγάλες εμπορικές αλυσίδες. Και από την άλλη, όλε όλο και περισσότερες εταιρείε και μικρές και μεγαλύτερες που εισάγουν πάρα πολλά αγαθά ε, μαζικής κατανάλωσης και κακής ποιότητος από την Κίνα. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει λοιπόν δεν άντεξαν. Δεν μου αρκεί ένα λεπτό κυρία Πρόεδρε για να μπω σε λεπτομέρειε, αλλά θα ήθελα να σα παρακαλέσω για το εξή. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τέτοιε εμπορικέ συμφωνίε και διαπραγματεύεται και συζητάει τέτοια πράγματα, τότε θα πρέπει να σκέφτεστε και τα συμφέροντα αυτών των μικρών ανθρώπων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θέλω να σας παρακαλέσω να μένετε εντός θέματος και να τηρείτε το χρόνο σας. Ο συνάδελφος Κούκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόθεση της αμοιβαίας συνεργασίας στην ε, Ασία είναι προς το συμφέρον όλων και γι' αυτό θέλω να στηρίξω τις διαπραγματεύσεις τις εμπορικές ανάμεσα στην Ένωση και την Ταϊβάν. Η σταθεροποίηση των σχέσεων ανάμεσα στην Ταϊβάν και την Κίνα κατέστησε δυνατή την επέκταση των ε, ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων στην Νοτιοανατολική Ασία και την Κίνα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερο τις ε, προόδους της Ταϊβάν στην έρευνα και στην ανάπτυξη ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και εμείς τις αντίστοιχές μας, τους αντίστοιχους μας τομείς. Η εμπειρία μας από τη Σλοβακία ναι ότι τέτοιου είδους εμπορικές σχέσεις προσθέτουν αξία. Θα πρέπει να προσβλέπουμε στις διαπραγματεύσεις για την προστασία των επενδύσεων και άλλες μορφές αμοιβαία αποφελών ε, συμφωνιών. Ευχαριστούμε κύριε Κούκανο, συνάδελφος Μπρόντζ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει με την Ταϊουάν εμπορικό έλλειμμα, αλλά πλεόνασμα στις υπηρεσίες. Το Ηνωμένο Βασίλειο έλλειμμα 3 προς 1 που υπονομεύει την βιομηχανία της Αγγλίας. Το πλεόνισμα στις υπηρεσίες μειώνεται κάθε χρόνο. Οι επενδύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου είναι 4 προς 1 των Ταϊβανέζων στο Ηνωμένο Βασίλειο χρηματοδοτείται έτσι ο ανταγωνισμός από την ε, Ταϊουάν. Η χώρα αυτή επενδύει σε οικονομίες ε, της Ασίας με χαμηλούς μισθούς. Ε, έχουν συνιστούν οι εισηγιστές διότι προωθεί τους στόχους του ΠΟΕ να υπάρξει, να ανοίξει το εμπόριο παγκόσμια διότι επιδιώκονται όχι στόχοι ευρωπαϊκοί, αλλά στόχοι παγκόσμιοι. Ο τελευταίος ομιλητής, ο συνάδελφος Μπίλαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ταϊβάν ε, είχε εκδηλώσει προθυμία να διαπραγματευτεί μια τέτοια συμφωνία επενδύσεων και εμπορικών σχέσεων. Ακόμα και δεν την έχουμε αναγνωρίσει ως ε, ανεξάρτητη χώρα, θα πρέπει να είναι προς το δικό μας συμφέρον μια τέτοια συμφωνία. Αλλά βέβαια να, δούμε και τη σχέση μας με το Πεκίνο, ε, και να μην ε, πέσουν αυτές στο βωμό της συμφωνίας με την Ταϊβάν. Αλλά τώρα φαίνεται ότι οι δύο χώρες έχουν έρθει πιο κοντά, μπορεί να μας βοηθήσει μια τέτοια συμφωνία, να έχουμε πρόσβαση στην αγορά και μπορεί να είναι εναλλακτική λύση και συμπλήρωση μια συμφωνίας με το Πεκίνο. Και επίσης ε, είναι δημοκρατικό το σύστημα κράτος δικαίου με πολυφωνία και πολυκομματισμό. Γι' αυτό είμαι υπέρ της εμβάθυνσης των σχέσεων με την Ταϊβάν και τα θέματα της προστασίας των επενδύσεων είναι πολύ σημαντικά και πολύ ευνοϊκά. Ιδιαίτερα σκεφτούμε πόσο ε, ανεπτυγμένη είναι η Ταϊβάν στις σύγχρονες τεχνολογίες. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος έχει το λόγο παρακαλώ κύριε Τεχάχτ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος διότι ήδη ανέπτυξα το θέμα σε σχέση με το, την προφορική ερώτηση στην εισήγησή μου. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας ε, ναι, φυσικά επί τη βάση του τι είναι καλύτερο από, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ευρωπαίους πολίτες. Για να τα πούμε ξεκάθαρα, δεν θα ε, διστάσουμε να προβούμε σε διαπραγματεύσει με την Ταϊβάν επειδή ίσω η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας δεν είναι κατά. Είναι δικό μας δικαίωμα, κυρίαρχο. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν άλλα κριτήρια που παίζουν ρόλο και αυτό είναι το δυναμικό ε, των διαπραγματεύσεων με την Ταϊβάν και σε σχέση με άλλες επιλογές. Θα πρέπει να πω ότι σε αυτή τη χρονική στιγμή όπου οι πόροι είναι εξαντλημένοι και λίγα λέω, δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιδέα του να γίνουν διαπραγματεύσει οι επενδυτικές συμφωνίες που θα καλύπτουν και την πρόσβαση στην αγορά και θα το εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο εν το χρόνο. Το λέω αυτό γιατί εκφράστηκε ομόφωνα στήριξη ε, υπέρ των στενών εμπορικών σχέσεων με την Ταϊβάν. Και σίγουρα θα επαναξετάσουμε το θέμα και στην Κομισιόν. Η συζήτηση έληξε. Το Προεδρείο έχει λάβει μία πρόταση ψηφίσματος και η σχετική ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.30 το πρωί. Και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη